Good afternoon, everybody. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινούμε με την απογευματινή μας συνεδρία. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ε, ε, εφαρμογή των ειρηνευτικών συμφωνιών του Μίνσκ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μακέιεφ, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής και Επικοινωνιών από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Αντρέας Χότμαν από το ειδικό αποστηλωμένο για την Ουκρανία, επικεφαλή τη ειδική ομάδα για την Ουκρανία από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Ραφαέλ Μακτίν Ντελαν. Λαγκάρτ, αναπληρωτή διευθυντή για τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Καλώ ήρθατε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω του ε, ε, καλεσμένου μα που βρήκαν τον χρόνο να έρθουν να μιλήσουν στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά ε, το ε, Μίνσκ ε, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ο τρόμος με τον οποίο η διαμάχη μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας θα επιληθεί και αυτό θα βοηθήσει όχι μονάχα τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά επηρεάζει και ολόκληρο το δυτικό κόσμο τα αίτια της αντιπαράθεσης δεν είναι πρόσφατα ε, είναι βαθιά ριζωμένα στα, στη σχέση μεταξύ της και Ρωσίας. Οι ε, διπλωματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ονορμανδίας έχουν επικεντρωθεί στο να αποτρέψουν την κλιμάκωση στρατιωτικής ε, διαμάχης ε, και την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, όμως ε, οι αριθμοί των θανάτων ε, ήδη από τον Ιανουάριο έχουν πεθάνει 45 άνθρωποι, ενώ 2016 έχουν τραυματιστεί και όλο αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς μια καλύτερη λύση για να σταματήσει η βία. Η συμφωνία του Μίνσκ ήταν μια, ένας δύσκολος συμβιβασμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ήταν ο μόνος ε, τρόπος ε, για αυτή, ε, σε αυτή τη φάση. Όμως δύο χρόνια μετά την υπογραφή του Μίνσκ είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για να αξιολογήσει σχετικά με το αν μπορεί να προσαρμοστεί στην πολιτική της για τη Ρουσία και την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί προσπαθεί περισσότερο στο να υποστηρίξει την Ουκρανία στις ε, μεταρρυθμίσεις της, να ενισχύσει ε, την σταθερότητα της χώρας. Ε, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Ουκρανίας, Γερμανίας και Γαλλίας να μας πούν σε ποια φάση της εφαρμογής βρισκόμαστε, το πώς μπορούμε εμείς ως κοινοβουλευτικοί να βοηθήσουμε στην διασφάλιση της κατάστασης ε, εάν θα πρέπει να έχουμε, πώς γίνεται να έχουμε μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός. Όλες αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις τις οποίες ε, οι συνάδελφοί μας θα θέλουν να σας θέσουν σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να δώσω το λόγο στον κύριο Αλέξη Μακέιεφ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ προς όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, για την ε, δέσμευσή τους και την υποστήριξή τους ε, προς την Ουκρανία και εμείς στην Ουκρανία το εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που ήρθατε σήμερα για να ακούσετε την έκθεσή μου αλλά και τις πληροφορίες των συνοδέλφων μου σχετικά με το τι συμβαίνει με το Μίνσκ και τη διαδικασία της Νορμανδίας, ε, τις διαπραγματεύσεις του Μίνσκ. Ε, την τελευταία φορά που ήμουν εδώ είχα τη τιμή να ενημερώσω αυτή την ε, επιτροπή τον Οκτώβριο πέρυσι περί τους 8 μήνες πριν και θα θυμάστε ίσως ότι είχα αναφέρει στοιχεία από το ε, μέτωπο, από την πρώτη γραμμή, τα οποία λαμβάνω τηλεφωνικά καθημερινά. Πρόκειται για στοιχεία ε, Ουκρανών άμαχων αλλά και ε, στρατιωτών οι οποίοι ε, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν καθώς επίσης και τα ονόματα αυτών. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορώ να σας φέρω καλά νέα. Η Ρωσία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση ε, να ε, τηρήσει το, ε, πιν, το Μίνσκ. Ο Πούτιν δεν κάνει τίποτα για να αποσυρθούν τα στρατεύματα από την Ουκρανία. Από τότε που συναντηθήκαμε δηλαδή πάνω από 200 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετές εκατοντάδες στρατιώτες αλλά και άμαχοι τραυματίστηκαν. Ε, ο αριθμός αυτός αυξάνεται και οι ε, ρωσικές ε, στρατιωτικές μονάδες αυξανόμενα επιτίθενται άμαχους. Οι Ουκρανοί έχουν πυροβοληθεί πάνω από 20.000 φορές το κατηλημένο Ντον ε, Πάσκ ε, λαμβάνει καθημερινά ε, όπλα από τη Ρωσία, κάτι το οποίο παραβιάζει το Μίνσκ, διατηρεί τις στρατιωτικές του μονάδες στην κατηλημένη περιοχή. Για να μπορέσουμε λοιπόν, ε, για να μπορέσουν να το γίνουν αυτό, η Ρωσία και οι υποστηρικτές της αντιτίθενται στην ε, εγκατάσταση της ε, μόνιμης αποστολής του ΟΑΣΕ στα σύνορα και μπορείτε να φανταστείτε ότι πρόκειται ε, για 400 ε, χιλιόμετρα ε, συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας τα οποία δεν ελέγχονται από την Ουκρανία. Οπότε λοιπόν υπάρχει τρομερή δυνατότητα για τους Ρώσους να φέρουν στρατιώτες, όπλα, παροχές. Όμως αυτό το οποίο κάνουν οι Ρώσοι είναι ότι προσπαθούν να διώξουν την αποστολή του ΑΣΕ και ίσως να ακούσατε ότι πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξαν ε, και οι πρώτες απώλειες ε, ε, όπου ένας, ένα μέλος του ΑΣΕ από τις Ηνωμένε Πολιτείε δολοφονήθηκε. Αυτό το οποίο κάνουν οι Ρώσοι από πέρσι το Φεβρουάριο είναι ότι όχι μόνο δεν πυροβολούν εναντίον υποδομών και, αλλά και άμαχους ενώ ταυτόχρονα καθημερινά ε, έχουμε τις ε, συναντήσεις ε, από τότε που έγιναν οι συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Νορμανδίας στο Μόναχο η Ρωσία έχει αναγνωρίσει μια σειρά παράνομων εγγράφων τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στον Τονβάς ε, τα οποία ε, παραβιάζουν τη συμφωνία του Μίνσκα. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Ρωσία είναι ότι η εγκαθιδρία ε, το ρουσικό ρούβλι ως νόμισμα στην περιοχή και με βίαιο τρόπο έχει λάβει υπό τον έλεγχό της όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή και ε, πέραν τούτου δεν βλέπουμε καμία πολιτική βούληση από την πλευρά της ε, Ρωσίας ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο του Μίνσκ και στο πλαίσιο της Νορμανδίας με τους ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν οδικό χάρτη για να μπορέσουμε να ε, βγούμε από, αυτό, ε, από αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο ε, απουσιάζει αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πολιτική βούληση. Από δική μας ε, πλευράς η Ουκρανία δεσμεύεται στην πλήρη εφαρμογή του ε, Μίνσκ. Ε, συνεργαζόμαστε με τους γερμανούς μας εταίρους και συντονίζουμε προσεκτικά όλες μας τις προσπάθειες προσπαθώντας να πείσουμε την Ρωσία αλλά και την ηγεσία της ώστε να αποτραβηχτεί και να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα απέναντι στην Ουκρανία μιλάμε για, την, για το κατελημένο Ντόν αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ε, το θέμα είναι η ε, Ρωσία να σταματήσει την παράνομη ε, κατάληψη της Κρυμαίας. Τώρα όσον αφορά το Ντόνμπας, ποιες είναι οι προσδοκίες μας σχετικά με την διεθνή κοινότητα, διότι σε αυτή τη φάση έχουμε μεγάλη ε, αλληλεγγύη από την πλευρά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατλαντικών μας εταίρων. Ε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επίσης βοηθά τους Ουκρανούς για να μπορέσει να λήξει αυτό το αιματοκύλισμα το οποίο ξεκίνησαν οι Ρώσοι. Αυτό το οποίο επιθυμούμε στον Τον Πάσκ είναι δηλαδή να υπάρξει μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει η διανομή βαρέων όπλων και ε, στρατιωτών στο ε, ελεγχόμενο ε, κομμάτι των Ουκρανικών σύνορων. Θέλουμε ο ΑΣΕ να λάβει πλήρη πρόσβαση στο κατεχόμενο Τον Πάσκ και να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των σύνορων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ε, να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα από ουκρανικό έδαφος και ταυτόχρονα να ε, ακολουθήσουν ε, διεθνή μέσα ασφαλείας. μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία πολιτικής λύσης παρά μόνο αν υπάρχουν τοπικές εκλογές στην περιοχή. Ε, το τελευταίο μου σχόλιο, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, είναι το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Και δεν υπάρχουν ε, πολλά εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο βασικό αυτών των εργαλείων είναι συνεχίσει με την πολιτική της μη αναγνώρισης για την παράνομη προσάρτηση της ε, Κρυμαίας και κανένα ε, δικαίωμα της Ρωσίας να ε, αναμειχθεί σε ε, εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας αλλά και τις κυρώσεις. Εκτιμούμε ιδιαίτερως τις αποφάσεις της Δευτέρας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις κυρώσεις για τη Ρωσία οι οποίες επεκτάθηκαν για ένα έτος και εκτιμούμε επίσης τις ε, οικονομικές ε, κυρώσεις οι οποίες ε, θα επεκταθούν στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήμασταν ευγνώμονες απέναντι στους ευρωβουλευτές αν υπερασπιζόσασταν την παράταση των κυρώσεων όχι για έξι μήνες αλλά για ένα χρόνο ε, το οποίο θα ήταν ένα πολύ σημαντικό ε, μήνυμα προς την ε, Ρωσία σχετικά με την ενότητα των συμμάχων μας αλλά και την υποστήριξη προς τους Ουκρανούς οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία τους και το δικαίωμά τους να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακέιεφ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντρέας Πρότμαν Οπότε τελικά θα αρχίσει ο κύριος ε, Ραφαήλ Μαρτίν Τελαγκάρτα να πληρωθεί διευθυντής για τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σα ευχαριστώ πολύ. Όντω με τον Γερμανό συνάδελφο Μπρότμαν μοιραστήκαμε κατά κάποιο τρόπο τα θέματα στις ε, παρεμβάσει μα. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω θυμίζοντα ε, κάποια διακυβεύματα τη Ουκρανική κρίση και να πω ότι αυτά τα διακυβεύματα καταρχάς αφορούν την Ουκρανία, όπως θύμισε και η Πρόεδρος και ο Ουκρανός συνάδελφος Μακιέφ, αυτή η ε, σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει ε, κοστίσει 10.000 θύματα και 20.000 τραυματίες. Σύμφωνα με τον είπα το αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται βοήθεια ανθρωπιστική επίγουσα σε αυτή τη χώρα που βρίσκεται στο ε, σπήλα της Ευρώπης. Θα χρειαστούν και ακόμα και αν σήμερα τελειώσει η κρίση, θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι ότου να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις. Σε δεύτερο διακύβευμα αφορά εμάς την Ευρώπη και τις σχέσεις μας με την Ουκρανία και ευρύτερα με τις γειτονικέ ανατολικές χώρε χώρες. Είναι πρόκληση για την ενότητα της Ευρώπης γιατί η Ρωσία είναι τμήμα της σύγκρουσης αλλά παραμένει και ένας ε, αδιαφεσβήτητος εταίρος μας. Γι' αυτό το λόγο η Γαλλία και η Γερμανία καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διαμεσολάβησης για να προσπαθήσουν να βρουν μια ε, πολιτική λύση τρίτη σειρά διακυβευμάτων είναι εν τέλει η αντικρουόμενες απόψεις που μπορεί να έχει κανείς για τις διεθνείς σχέσεις. Από τη μια πλευρά έχουμε μια πολιτική που βασίζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της πολυμερικότητας της πολιτικής που μας εμπνέει και από την άλλη πλευρά μιας πολιτικής ισχύω και ζωνών επιρροής που ευνοεί την, το μέγεθος ακόμα και με τίμημα την απομόνωση. Τώρα, να σας, να σας πω που βρισκόμαστε στη διαδικασία. Εγώ παρενέβην όντω και είχα την ε, τύχη να είμαι προσκεκλημένος τον Οκτώβριο του 2015 με τον κύριο Μοκίγεφε και τον ε, τότε γερμανό μου συνάδελφο και σας είχαμε ενημερώσει για τις διαμεσολαβητικές μας εργασίες για την εφαρμογή του Μίνσκ, συνεργασία γαλλογερμανική και τι κάναμε έκτοτε. Είχαμε διάφορες διαδοχικές ε, συσκέψεις ε, ξεκινώντας με μία διάσκεψη κορυφής στις 19 Οκτωβρίου στο Βερολίνο ε, του 19 Οκτωβρίου του 2016 τη διαδικασία τύπου Νορμανδίας. Έκτοτε έγιναν δύο συσκέψεις υπουργικού επίπεδου πάλι υπό τη μορφή τύπου Νορμανδίας η μία στο Μίνσκ και η άλλη στο 17 Φεβρουαρίου στο Μόναχο. Στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορες συνεδριάσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, κυρίως των διπλωματικών ε, συμβούλων ή των αναπληρωτών του, του Προέδρου και της Καγκελαρίου. Η τελευταία εξ αυτών έλαβε χώρα το στις 6 Απριλίου ε, στο Μίνσκα ε, έχουν γίνει και ε, διπουργικές ε, συσκέψεις σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών. Είναι οι πολιτικοί διευθυντές και οι υφυπουργοί των Υπουργείων μας με τριμερείς ομάδες επαφών του ΟΑΣΕ. Δηλαδή ειδική εκπρόσωπος του Προέδρου της ΟΑΣΕ και τέσσερις συντονιστές των ομάδων εργασίας. Στόχος αυτών των συσκέψεων είναι να υπάρξει επαφή ανάμεσα στις συνεδριάσεις τύπου Νορμανδίας και τις τύπου τριμερού που κάθε δύο εβδομάδε στο ΜΕΝΣ ασχολούνται με πολιτικά θέματα, θέματα ασφαλεία, ανθρωπιστικά και οικονομικά ζητήματα. Τι έχουμε καταφέρει με όλα αυτά. Θα σα πω δύο λόγια για την πολιτική διάσταση των συμφωνιών του ΜΕΣ και την εφαρμογή του και την ανθρωπιστική πτυχή και μετά θα δώσω το λόγο στον Γερμανό συνάδελφο όσον αφορά τι πτυχέ ασφάλεια και τι οικονομικέ πτυχέ. Στον ε, πολιτικό τομέα, Έχουμε τέσσερα σύνολα. Το πρώτο αφορά την συνταγματική μεταρρύθμιση που αφορά την αποκέντρωση, δηλαδή ε, εκεί όπου έχουμε κάποια περισσότερα αποτελέσματα γιατί υπάρχει ένα σχέδιο συνταγματικής μεταρρύθμισης που εγκρίθηκε από τη Ράντα σε πρώτη ανάγνωση τον Αυγούστο του 2015. Ε, τώρα, για το ειδικό καθεστώς για ορισμένες ε, ε, ε, περιοχές όπως το Ντούνμπας. Τον περασμένο Οκτώβριο στη διάσκεψη κορυφής του Βερολίνου δεν καταλήξουμε, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε υπό τον τύπο της Νορμανδίας και υπό τον τύπο Σταν Μάγερ όπως αποκαλείται, δηλαδή μέσω μιας διαδικασίας που είχαμε επεξεργαστεί ένα χρόνο νωρίτερα στις 2 Οκτωβρίου 2015 στο Παρίσι και έτσι εκεί εξηγούμε πώς θα εφαρμοστούν τα διάφορα πολιτικά στοιχεία των συμφωνιών του Μίνσκ. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει η αρχή από έναν εκλογικό νόμο για τις τοπικές εκλογές στο Ντόμπας, πράγμα που πρέπει να εγκριθεί από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο με μια προπαρασκευαστική φάση για τις εκλογές που απαιτεί την ύπαρξη ασφάλειας. Έπειτα ε, θα γίνει η ενέργεια εκλογών και τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί εκλογές, το ειδικό καθεστώς αυτών των εδαφών θα χορηγηθεί και θα αρχίσει να ισχύει ε, προσωρινώς και στη συνέχεια την ημέρα που ο ΑΣΕ και το Διεθνές Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΣΕ που θα κρίνει μέσω αποστολής ε, εμπειρογνωμόνων ότι έγιναν εκλογές όπως ε, δει, δηλαδή σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια, τότε το καθεστώς αυτό θα οριστικοποιηθεί. Τελευταίο στοιχείο είναι ότι την επομένη, την επαύρη των εκλογών, ε, ο νόμος περί αμνηστίας που υιοθετήθηκε από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2014 που δεν έχει ισχύσει, θα άρχιζε να ισχύει. Αυτή είναι η λιλουχία, την οποία θυμήσαμε και επιβεβαιώσαμε στο διάσκεψη κορυφής του Βερολίνου στις 19 Οκτωβρίου και επ' αυτόν εργαζόμαστε. Για να προχωρήσουμε ακριβώ ε, να σα πω ότι εργαζόμαστε και επί μια διαδικασία για τι τοπικέ εκλογέ. Πώ δηλαδή θα διενεργηθούν αυτέ οι εκλογέ στον Ντόν εδώ έχουμε επαφές σε τριμερούς τύπου ομάδων εργασίας για τα πολιτικά ζητήματα που συνεδριάζουν στο ΜΙΣ κάθε δύο εβδομάδες, αλλά φυσικά με τη στήριξη της ε, ε, διαπραγμάτευση τύπου Νορμανδίας. Και για τον νόμο περί θα πρέπει αυτός να αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με τον τύπο Σταν Μάγερ. Υπάρχει ήδη η νομοθεσία αυτή, έχει εγκριθεί από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2014. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο διάλογος που προβλέπεται από τις συμφωνίες του Μίνσκ έχει ξεκινήσει για καθένα από τα μέτρα της πολιτικής ε, πτυχής. Η Ουκρανία έχει συμμετάσχει και έχει αναλάβει δεσμεύσεις. Ωστόσο, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι για να προχωρήσει η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διάστασης θα πρέπει να γίνουν και προόδοι στα θέματα ασφάλεια. Τα δύο αυτά πάνε χέρι-χέρι. Αυτή είναι η φιλοσοφία των συμφωνιών του ΜΙΣ και ότι μάλιστα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ασφάλεια και από μια πραγματική πάυση του πυρός, μια πραγματική ανακοχή ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε στα πολιτικά θέματα. Και γι' αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε παράλληλα στις δύο αυτές πτυχές που είναι ουσιώδεις για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. τώρα, η άλλη πτυχή είναι η ανθρωπιστική, που φυσικά έχει και αυτή μεγάλη σημασία και που συζητώνται επίσης πάλι στο στην, υπό τη μορφή της τριμερούς ομάδας επαφής ε, που ε, προβλέπεται από το Μίνσκ, από τη συμφωνία του Μίνσκ ε, και με εμπειρογνώμονες από την ΟΑΣΕ και εργαζόμαστε και προσπαθούμε να στηρίξουμε με πολιτικό τρόπο μέσω της διαδικασίας τύπου Νορμανδίας. Πρώτον, ανταλλαγή κρατουμένων. Σημαντική κόεργο έχει γίνει από το 2015. Τα νούμερα μπορεί να ποικίλουν, αλλά υπολογίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 180 με 200 κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν από το 2015. Παραμένουν ακόμα αρκετοί και από τις δύο πλευρές και εργαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Και εκεί δηλαδή η, ομα... η τριμερής ομάδα εργασία εργάζεται επί όλων των τεχνικών ε, πτυχών όσον αφορά την αναγνώριση, ταυτοποίηση κτλ. Και εμείς ε, υπό τη διαδικασία Νορμανδίας, δηλαδή σε επίπεδο αρχηγών κρατών, προσπαθούμε να δώσουμε πολιτική στήριξη ώστε να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή. Ε, συνεχίζεται η δουλειά από αυτών των θεμάτων. Δουλεύουμε επίσης για τους αγνοούμενους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα ανθρωπιστικά θέματα και στο πλαίσιο της ε, και σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Επίσης, ε, ε, δυστυχώς για τον Τόμπας η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη όταν έχουμε συνεδριάσει σε πολιτικό επίπεδο επιμένουμε πολύ ε, όσον αφορά τη Ρωσία. Επιμένουμε προς τη Ρωσία να ζητήσει από τους ε, ε, ε, ε αποσχιστές να, να, να επιτρέψουν την διέλευση των ανθρωπιστικών της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάτι ακόμα, για να επιτραπεί η ανταλλαγή ανθρώπων ανάμεσα στις δύο πλευρές ε, του μετόπου, και αυτό είναι κάτι που το επιμένουμε καθημερινά, υπάρχει μια κάπως ατυχή διαδικασία, ατυχής διαδικασία συνοριοποίησης όλης της γραμμής του μετόπου, όπου βλέπουμε να μειώνονται οι, οι συναλλαγές και κυρίως οι οικονομικές συναλλαγέ. Προσπαθούμε λοιπόν να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις ανθρώπων από τα φυλάκια, στηρίζοντας τα αιτήματα των εν λόγω ανθρώπων και στηρίζοντας τις προσπάθειες της Ουκρανικής πλευράς ώστε να ελαφρυνθεί η διαδικασία για αναγνώριση των ανθρώπων αυτών, να μπορέσουν επίσης να μεταφέρουν ας πούμε, πιο μεγάλες ποσότητες προϊόντων, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ε, μεταφορές ε, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι κάποια θετικά στοιχεία, γίνεται κάποια πρόοδος, υπάρχει μια κάποια διευκόλυνση στις συναλλαγές. Για τον αριθμό των φυλακίων που είναι ανοιχτά είναι αρκετά περιορισμένος και εξαρτάται φυσικά από την ασφάλεια γιατί τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δυσχεροί. Μόνο ένα σημείο υπάρχει ανοιχτό για, την, ε, για το Dance και μάλιστα η διέλευση δεν είναι πάντα εύκολη και στο Ντονιέξκ υπάρχουν τρία σημεία διέλευσης. Το ένα είναι κλειστό ε, στο η τοποθεσία Ζόλοτε και κάνουμε έκκληση προς τις δύο πλευρές να καταβάλουν προσπάθειες να ανοίξει αυτό το σημείο διέλευσης για να διευκολυνθούν και οι άνθρωποι που ζουν εκεί και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Και από την ανθρωπιστική άποψη αυτό που κάνουμε επίσης είναι ότι στηρίζουμε από πολιτικής άποψης προσπάθειες που στόχο έχουν την αποναρκοθέτηση Πολύ σημαντικό επίσης θέμα. Υπάρχουν ε, θάνατοι αμάχων που οφείλονται στις νάρκες. Μάλιστα θύμα έπεσε και ένα μέλος της αποστολής του, του, του ΟΑΣΕ. Θύμα νάρκης δηλαδή καλούμε τα εμπόλεμα μέρη, γιατί αυτοί φέρουν την πρώτη ευθύνη, εκείνοι έχουν αρκοθετήσει όλη την περιοχή. Προσπαθούμε βέβαια να τους βοηθήσουμε και να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία. Αυτά λοιπόν από ανθρωπιστική άποψη και τώρα να δώσω το λόγο στον Γερμανό μου συνάδελφο για την ασφάλεια που είναι πολύ σημαντική βεβαίως και για όλα τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ανδρέας Μπρότμαν επικεφαλής της Task Force ε, για την Ουκρανία ε, του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ε, έχετε 10 λεπτά παρακαλώ. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Ραφαέλ που ξεκίνησες με την έκθεσή μας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα ζητήματα ασφαλείας, στα οικονομικά ζητήματα και να κλείσω με κάποια σχόλια για τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Κατά τη γνώμη μας, το πιο επίγον ζήτημα στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ είναι να βελτιωθεί η κατάσταση σε επίπεδο ασφαλείας ε, στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν η Γερμανία και η Γαλλία προσπαθούν να δώσουν μια νέα όθηση στη διαδικασία του Μίνσκ. Επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Αυτό ήταν και στην καρδιά ε, της συνάντησης ε, που έγινε σε επίπεδο αναπληρωματικών ε, υπουργών εξωτερικών, ε, υπουργών εξωτερικών που χώρα στο Βερολίνο στις 30 ε, Μαΐου. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις εκθέσεις των ειδικών αντιπροσώπων της ΟΑΣΕ, του πρέσβη Ζάιντι, Ζάιντι και τους εκπροσώπους των ομάδων εργασίας της τριμερής ομάδας επαφής προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία ε, Μίνσκ και τις σχέσεις με το ε, format Normandy. Ε, θέλουμε να επανέλθουμε στην αρχική λογική της συμφωνίας του Μίνσκ, σύμφωνα με την οποία μια σταθερή κατάσταση σε επίπεδο ασφάλειας είναι εκ των ουκ άνευ για όλα τα λοιπά βήματα, ιδιαίτερα τα πολιτικά βήματα. Τρία ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά εδώ. Πρώτον, μία εχεκυρία η οποία να είναι αξιόπιστη, να, δεύτερον ε, να αποσυρθούν τα βαρέα όπλα και τρίτον να υπάρξει αποδέσμευση. Ε, στις 4 Απριλίου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το θέμα της ασφάλειας. Αποφασίστηκε ότι η δέσμευση για γεχηρία που είχε θεσπιστεί πριν, τα, πριν το Πάσχα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Έτσι λοιπόν οι τέσσερις ηγέτες του Νόρμαντι ε, ενίσχυσαν την εκεχειρία του Πάσχα σε μια τηλεφωνική συνομιλία και σε μια κοινή δήλωση που ακολούθησε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε την εκ νέου δέσμευση στην Νόρμαντι ε, για να γίνει μια συνεδρίαση και η συζήτηση επιτόπου παραμένει εξαιρετικά ε, ταραγμένη. Έχουμε και σημαντικό αριθμό θυμάτων ε, πολιτών, διότι βομβαρδίζονται ε, κατοικημένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο ε, πλήττει και τις διάφορες υποδομές, ε, ε, για τη διαχείριση λιμάτων γενικότερα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένε δράσεις και πιο συγκεκριμένα πρέπει να αποσυρθούν τα βαρέα όπλα. Έχει ζητηθεί να λάβουμε κάποιε πληροφορίες σε ό,τι αφορά αυτό το βαρύ οπλισμό. Ελπίζουμε ότι θα δοθεί συνέχεια σε αυτό το αίτημα. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η ασφάλεια της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ. Είχαμε ένα φωνικό συμβάν στις 24 Απριλίου ε, ένας Αμερικανός ε, ε, γιατρός που συμμετέχει σε αυτήν την αποστολή καθώς και ένας Τσέχος και ένας Γερμανός εκπρόσωπος τραυματίστηκαν ο Αμερικανός έχασε τη ζωή του ε, είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να γίνει μια έρευνα για το συμβάν αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόσβαση στο σημείο όπου συνέβη ε, το περιστατικό είναι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκο, Λουγκάνσκο αυτό που καλούνται δηλαδή εκεί που βρίσκονται οι αποσχιστές, οι αποσχιστικές δυνάμεις. Ε, λόγω αυτού του συμβάντος στις 23 Απριλίου έχουμε δει ότι υπάρχει μείωση της δυνατότητας της αποστολής να παρακολουθεί, να εποπτεύει την κατάσταση, διότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Και βεβαίως ε, η αποστολή βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, υπό συνεχή παρενόχληση και επιθέσεις από την πλευρά των αποσχιστών. Ως αποτέλεσμα αυτής της, αυτού του συμβάντος, στις 23 Απριλίου, πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα ε, η αφαίρεση των ναρκών πρέπει να αρχίσει τουλάχιστον άμεσα η καταγραφή των ναρκοπαιδείων ε, έχει ζητηθεί από τον πρέσβη Απακάν ε, έχουν ζητηθεί χάρτες ε, σε ό,τι αφορά τις ναρκοθετημένες περιοχές θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε αυτούς τους χάρτες σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα τα οποία εξετάζονται και στην, επίπεδο του Normandy 4 αλλά και στο οικονομικό επίπεδο τρία ζητήματα εδώ στις συζητήσεις. Πρώτον, υπάρχουν τάσεις διάλυσης στον Ντόμπας. Δεύτερον, το θέμα της αντωνευοδευμού σε νερό. Και τρίτον, τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά. Η Γαλλία και η Γερμανία ανησυχούν ιδιαίτερα για την, ε, τις τάσεις, τις διαλυτικές ε, στην Ντόμπας, στον Ντόμπας είναι κάτι που υπονομεύει την παράγραφο 8 του πακέτου μέτρων του Μίνσκ που αναφέρει ότι οι οικονομικές, ε, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ και των δύο πλευρών του Ντόμπας πρέπει να διατηρηθούν. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μονομερών μέτρων από την αρχή του έτους που δυστυχώς οδήγησε σε μια ε, λογική αντιπίνων όπου κάποιος μπλοκάρει στις δρομικές ε, ε, γραμμές οι Ουκρανοί ακτιβιστές και αυτό οδήγησε σε απαλωτρίωση επιχειρήσεων Ουκρανικών από την άλλη πλευρά και η Ρωσία δεν βοήθησε βέβαια διότι εξέδωσε ένα διάταγμα που αναγνωρίζει έγραφα των αποσχιστικών δυνάμεων και των, ε, το αποκαλούμενων δημοκρατιών ε, και τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ουκρανίας τον Μάρτιο αποφάσισε να ξεκινήσει επίσημο μπλόκο στα προϊόντα ε, που, που κατευθύνονται προς τις περιοχές αυτές. Στο Βερολίνο στις 30 Μαΐου Προσπαθήσαμε να υποβάλουμε μια πρόταση, η Γερμανία και η Γαλλία, ε, για το πώς ε, αυτή η ατυχής, εξαιρετικά ατυχής κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Η βασική ιδέα είναι να έχουμε ταυτόχρονη απόσυρση των μέτρων και της απαλωτρίασης από την πλευρά των αποσχεστικών δυνάμεων και από την πλευρά του ε, μπλόκου που υπάρχει στη μεταφορά προϊόντων από την άλλη πλευρά. Ε, τώρα το θέμα του εφοδιασμού ε, σε νερό από τις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση υπάρχει διαφορά μεταξύ Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Εδώ, στην πλευρά του Λουγκάνσκ, υπάρχουν ζητήματα πληρωμών. Πληρωμή, δηλαδή, από την πλευρά των προσχεστικών δυνάμεων προς τους παρόχους ύδατος, προς την ε, πλευρά την κυβερνητική χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αξιόπιστο και βιώσιμο για την πληρωμή για την ώρα η πληρωμή λαμβάνει χώρα σε ρευστό ε, με σε, σε μία ασφαλής οδούς στο Λουγκάνσκ χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ε, πληρωμής που να μην βασίζεται στα ρευστά Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τι περιοχέ που ελέγχονται από τι αυτοπροκαλούμενε λαϊκέ δημοκρατίε, ε, υπάρχει πιο πολύ θέμα ασφαλεία στον ανεφορισμό του νερού. Είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα. Ε, οι ε, διάφοροι σταθμοί ε, συγκέντρωσης νερού συχνά βομβαρδίζονται. έπρεπε λοιπόν να επισκευαστούν από προσωπικό που κάνει μια ηρωική δουλειά σε σύντομες, σύντομα χρονικά διαστήματα και χειρίας. Υπάρχει τώρα βέβαια η ανησυχία ότι τώρα με το καλοκαίρι και τη ζέστη το πόσιμο νερό ε, αρχίζει να ε, μην είναι πια στην κατάλληλη κατάσταση, να μην έχει την κατάλληλη ποιότητα. Ε, γενικότερα υπάρχει ένα θέμα περιβαλλοντικό στην περιοχή. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια αξιολόγηση της κατάστασης με το νερό, ε, ιδιαίτερα με τις, ε, τα ορυχεία τα οποία έχουν πλημμυρίσει στην περιοχή. Στην ομάδα εργασίας έχουμε προτείνει να δημιουργηθεί μια ομάδα πυρογνώμων για να εξετάσει την κατάσταση των ορυχείων και από τις δύο πλευρές ε, δυστυχώς οι αποσχιστικές δυνάμεις από το Λουγκάνσκ δεν έχουν συμφωνήσει για να συμβεί αυτό. Κάποια σύντομα σχόλια για το πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Ελπίζω να μην ήταν πολύ μαύρη εικόνα που σας περιγράψαμε, εγώ και ο συνάδελφος. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα θέλαμε μια πιο ουσιαστική πρόοδο ε, κατά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Όμως η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να είναι αποφασισμένες ε, και γι' αυτό σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε σημεία επαφή υψηλού επίπεδου πριν το καλοκαίρι. Το επόμενο βήμα θα είναι και μια να καλέσουμε μια διάσκεψη των τεσσάρων ηγετών του Normandy 4 ε, στα τέλη Ιουνίου και με τον νέο Γάλλο πρόεδρο ελπίζουμε ότι θα δοθεί έτσι μια νέα όθηση στην όλη διαδικασία Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί. Uh, uh, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τους ομιλητές για τις δηλώσεις και τις παρουσιάσεις τους και τώρα το λόγο έχουν τα μέλη μας. Τέσσερα άτομα έχουν στήσει το λόγο. Ζητήστε το λόγο για να μοιράσουμε και το χρόνο. Ο κύριος Τέτινα πρώτα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ε, καλωσορίζω εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν ε, με ενδιαφέρει ποιος θα απαντήσει την ερώτηση, απευθύνεται σε όλους. πρώτον, σκεφτόμασταν ότι ε, τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση της Μαριούπολης ότι ε, ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια. Ε, έχουμε ακόμα ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν εκεί πέρα και οι συμφωνίες του Μίνσκ είχαν ως στόχο τους να ε, διατηρηθούν οι κυρώσει απέναντι στην ε, ε, Ρωσία. Όμως κατά τα άλλα δεν λειτουργούν καθόλου. Οι ίδιοι αναφέρατε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, συνεχίζονται οι μάχες. Έτσι λοιπόν το ερώτημά μου είναι υπάρχει ένα σχέδιο Β ένα σχέδιο το οποίο πράγματι θα μπορούσε να λήξει τον πόλεμο ε, θα μπορούσε η δυνατότητα ε, να δώσουμε όπλα ε, στην Ουκρανία, αυτές τις οποίες χρησιμοποιεί και ο αντίπαλος, αλλά δεν έχει στη διάθεση της η Ουκρανία. Υπάρχει λοιπόν σχέδιο Β για το Μίνσκ και το άλλο ερώτημα αφορά τις εκλογές. Όταν τελευταία φορά βρέθηκα στην περιοχή, ο κυβερνήτης Τσιμπρίτσκι μου είχε πει ξεκάθαρα ότι η Γαλλία και η, και η Γερμανία πιέζει να γίνουν περιφερειακές εκλογές στην περιοχή και μας είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να οργανώσουμε εκλογές σε μια κατάσταση όπου στους δρόμους υπάρχουν ε, τάγκ. Ε, δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο ε, μαζί. Και σας ρωτώ, λοιπόν, η Γερμανία και η Γαλλία σκοπεύουν να ε, επιμείνουν ε, στο να υπάρξουν εκλογές όταν θα υπάρχουν ε, εχθρικές εκλογές ή θέλετε να γίνουν εκλογές εδώ και τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στέτινα. Ακολουθεί ο κύριος Τεσπάκερ και παρακαλώ τηρήστε το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ε, μου δόθηκαν απαντήσεις ε, στα ερωτήματα τα οποία είχα καθώς ερχόμουν εδώ. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, όσοι έχετε βρεθεί εκεί πέρα, ε, δεν υπάρχει τίποτα το καινούργιο ακόμα. Ε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, η οποία επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Είναι επικίνδυνη για τους ε, άμαχους ε, και είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ακόμα έναν, ένα μεγάλο πονοπάτι να διανύμουμε. Όμως χαιρετίζω την Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες προσπαθούν να αναβιώσουν το Μίνσκ, το οποίο είναι το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το οποίο επικεντρώνεται ε, στην ασφάλεια ε, και τη σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης από την πλευρά της Ουκρανίας ε, υπάρχουν πολλά να γίνουν. Το συνταγματικό πλαίσιο για ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Όμως έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με την εκαθάριση των αρκών. προσπαθήσαμε, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ε, ε, ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διεθνής βοήθεια από χώρες που έχουν ειδίκευση πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι η δική μου χώρα έχει ε, μια ειδικότητα πάνω σε αυτό. κάποια κράτη-μέλη ίσως θα μπορούσαν να παρέμβουν και να βοηθήσουν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε προετοιμασμένοι να σκεφτούμε ε, το επόμενο βήμα που θα γίνει. Η περιοχή του Ντονπάς ε, νομίζω ότι θα χρειαστεί ε, υποστήριξη, πρακτική υποστήριξη από από εμάς. Ελπίζω να έχουμε κάποια επιτυχία ούτως ώστε να μπορέσουμε να επανενσωματώσουμε την περιοχή στην Ουκρανία αλλά και στην ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα ο επόμενος ομιλητής, ε, ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε. Είναι σημαντικό να ακούσουμε όχι μόνο από μία χώρα, αλλά και από τους ε, Ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν στο Μίνσκ. Είναι ένα παράδειγμα υβριδικού πολέμου ε, είναι κάτι το οποίο ε, είχε ξεκινήσει η Ρωσία ήδη από το 1970. Από το 1917 θα πρέπει να εξετάσουμε την πρόσφατη κατάσταση με τους ε, Ουκρανούς επιχειρηματίες οι οποίοι έπεφταν θύματα συμμοριών στις περιοχές. Ε, είναι αυτό λοιπόν ένα ε, ζήτημα ε, στο, για τη συζητήση στο πλαίσιο του Μίνσκ και κάτι ακόμα. Ο συνάδελφός μου, κύριος Στέτοβα, ρώτησε κάποιες εναλλακτικές για το Μίνσκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, ο Τίλορσον είχε ε, πει ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις και εκτός του πλαισίου Μίνσκ. Ε, πώς πιστεύετε ότι σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα ε, του Υπουργού των ΗΠΑ. Και όσο λοιπόν οι διπλωμάτες της Γαλλίας και της Γερμανίας ε, θεωρούν ότι θα πρέπει στην διμερή διάταξη να υπάρχει το Μίνσκ και η Ουκρανία, αυτό υπάρχει και ακολουθεί η κυρία Χόμπς. θα ήθελα σε ένα γενικότερο ε, πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και η Γερμανία διαπραγματεύονται να αντιμετωπίσουν τις συμφωνίες του Μίνσκ ως ε, μια ε, συμφωνία όπου θα πρέπει να επιτευχθούν τα σημεία αυτών των συμφωνιών ή ταυτόχρονα βλέπουν και το ζήτημα της ε, κατοχής ε, και του πολέμου, το οποίο είναι μια εξέλιξη που αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι κατά την άγνώμη μου, ε, στο πλαίσιο αυτής της ενόχλησης για την μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων, ξεχνάμε το μεγαλύτερο πλαίσιο όπου αυτός ο υβριδικός πόλεμος αποτελεί ένα κίνδυνο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι λοιπόν χάνουμε ε, αυτή την εικόνα ε, και με την όλη συζήτηση που γίνεται και για το ΝΑΤΟ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι ε, κάθονται και συζητούν για τις κυρώσεις και για το αν θα γίνουν εκλογές στο Λουκάντσκ ή εάν θα αποτραβηχθούν τα τάγκς ή όχι και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπιστεί ε, τα συμφέροντά της. Και ε, μέσα σε αυτό το ερώτημα θα με ενδιαφέρει επίσης ε, να μου αναφέρετε αν προσπαθείτε να σχεδιάσετε πώς θα ήταν μια ε, απόσυρση των ε, στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές, αν στη συνέχεια ε, σχεδιάσετε σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο. Αν φτάναμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια πώς θα διασφαλίζονταν τα σύνορα και από ποιον. Ευχαριστούμε και τώρα έχουμε τρεις ακόμα που ζήτησαν ε, τρεις ομιλητές ε, και ε, αν μπορείτε να είστε όμως σύντομοι, 1,5 λεπτό συνολικά. Κυρία Πρόεδρε. να μην προσμετρηθεί αυτή η εισαγωγή μου στο 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, ε, πληροφορίες ε, που μας δώσατε, όμως έχοντας ακούσει όλα τα σχόλια σχετικά με την εφαρμογή ή μάλλον τη μη εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ μου δίνεται η αίσθηση ότι η ε, πέραν από την μια κάποια κατάδοση του, του ε, πυρός ε, δεν υπάρχει καμία άλλη εφαρμογή. Αυτή η παράλογη ιδέα ότι θα γίνουν εκλογές με στρατιωτική παρουσία αυτό το ζήτημα για ειδικό στάτους, αυτή η κλιμάκωση που γίνεται και ε, το ε, γεγονός ότι ε, δεν, γίνεται ανταλλαγή, δεν γίνεται ομήρων, αγνοουμένων, όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για μια παγωμένη διαμάχη. Είμαι πολύ αισιόδοξοι ή απεσιόδοξη. Υπάρχουν καθόλου αισιόδοξε ειδήσει όσον αφορά τι συμφωνίε του Μίνσκ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η δική μου αίσθηση είναι πως οι κυρώσεις βρίσκονται ε, σε επίπεδο που όλοι τις αγνοούν. Και το ερώτημα μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία εφαρμογή ε, των συμφωνιών του Μίνσκ. Ίσως ε, θα ήταν χρήσιμο αν είχαμε πολιτική βούληση για να σκεφτούμε να αυξήσουμε και να επεκτείνουμε τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καλνιέτε. Η κυρία Πιτέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στις διάφορες πτυχές της κατάστασης στην Ουκρανία. Είναι πολλά τα ζητήματα, όμως ε, το ερώτημά μου εμένα είναι το εξής. Μήπως θα μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει αλλάξει τελικά από την περασμένη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό πριν από μερικού μήνε. Μπορείτε με συγκεκριμένο τρόπο, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο, να μα πείτε ποια πρόοδο έχει σημειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Αντρικέ είναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις παρουσιάσεις. Ήθελα να πω ότι εξετάζοντας από κοντά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και γύρω από την Ουκρανία, έχω την εντύπωση ότι η εφαρμογή, η μη εφαρμογή της, της συμφωνίας του Μίνσκ έχει οδηγήσει αυτό το πάγωμα, σε αυτό το αδιέξοδο. Το έχουμε δει αυτό και στη Μολδαβία και στη Γεωργία και είναι πραγματικά λυπηρό. Το ρεύμα μου είναι προς τον κύριο Μακέγεφ, ε, συγγνώμη, θα επαναλάβω αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος. αυτή η θέση των Αμερικανών. Πριν από μερικούς μήνες ακούσαμε από τη Washington ότι υποστηρίζουν 100% την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Αναφέρονται σε κάποια νέα μορφή προσέγγισης για να βρεθεί λύση. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό. Ευχαριστώ και τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να κατανείμετε το χρόνο που θέλετε εσείς. Έχει τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ποιος θα ξεκινήσει. Ναι, καλύτερα να αρχίσω εγώ. Θα με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι βέβαια, διότι σίγουρα θα πρέπει να ακυρώσω και το δείπνο και το βρενό πρωινό αν είναι να απαντήσω όλα τα ερωτήματα και δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Σας ευχαριστώ πάντως για τα ερωτήματα. Από τα ερωτήματα αυτά προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη ε, εκ μέρου σας για να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Οι κυρώσεις δεν λειτουργούν. Ακούστε, λειτουργούν οι κυρώσεις. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Οι κυρώσεις λειτουργούν διότι η Ρωσική Ομοσπονδία από κοινού με, με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου ε, υποφέρει. Υποφέρουν οι Ρώσοι. Δεν το παραδέχονται, αλλά υποφέρουν. Εν ώψη λοιπόν ε, των, της προεδρικής εκλογής το 2018 ε, στη Ρωσία ε, θα καταλάβουν τι συμβαίνει ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχει αυτή η προπαγάνδα που τους, έχει, που τους κάνει πλήση εγκεφάλου αλλά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στο Κρεμλίνο. Σίγουρα υποφέρουν από τις κυρώσεις αυτές. Τώρα πρέπει να πω κύριε Στετίνα ότι αποκοινούμε με τη Γερμανία και τη Γαλλία ε, εργαζόμαστε χέρι-χέρι. Δεν υπάρχει κάποια πίεση δηλαδή. Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ηγετών μας. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Με τον νέο Γάλλο πρόεδρο ενδεχομένως ε, ε, θα έχουμε μια σημαντική όθηση στην όλη διαδικασία ο πρόεδρος μας θα συναντήσει σύντομα τον πρόεδρο της Γαλλίας σε ό,τι αφορά το ρόλο των ΗΠΑ. Σε δύο ώρες ο πρόεδρος μας, ο κ. Ποροσέγκο, θα συναντήσει τον κύριο Τραμπ στις ΗΠΑ. Οπότε σίγουρα θα έχουμε νέα στοιχεία από τη Βόσιγκτον. Πάντως είναι σημαντικό να πούμε ότι οι ΗΠΑ πάντα υποστήριζαν ε, τη Γερμανία και τη Γαλλία και το συντονισμό αυτό, το συντονιστικό, αυτό μηχανισμό. Ε, έχουμε ακούσει από τη Βόσινγκτον από τότε που ανέλαβε ο κύριος Τραμπ, ε, έχουμε ακούσει μόνο υποστήριξη ε, στην Ουκρανία. Δεν θα υπάρξει συμφωνία πίσω την πλάτη της Ουκρανίας. Θα ακολουθήσουμε τη λογική της συμφωνίας του Μίνσκ ε, εκεχηρία και πολιτική λύση. Αυτό λέει η συμφωνία. Η εκεχηρία όμως δεν λειτουργεί. Είναι υβριδική η εκεχηρία, έτσι. Είναι κάτι που έχουν, ε, ε, έχουν εφεύρει οι Ρώσοι. Δεν το κάνουν μόνο στην Ουκρανία, το κάνουν και στη Συρία. Ε, δηλαδή αποφασίζουν εκεχηρία και την επόμενη μέρα ε, την παραβιάζουν. Έχει κάποια υβριδικά στοιχεία όπως καταλαβαίνετε. η ρωσική στάση, όπως με την εκεχηρία. Συζητήσαμε βεβαίως ε, το θέμα ε, της ε, απαλωτρίωσης ε, των ουκρανικών επιχειρήσεων. συζητήθηκε στην ομάδα του Μίνσκ, προτάθηκε από τη γερμανική και τη γαλλική πλευρά ένα δρόμο για να, να βρεθεί μια λύση. Οι Ρώσοι δηλαδή να αποσύρουν αυτές τις αποφάσεις, να επιστρέψουν αυτήν την ιδιοκτησία τους κατοχούς της. Ευχαριστώ κυρία Καλνιέτε που αναφερθήκατε στο ζήτημα των εκλογών και εσείς κυρία Στετίνα. Όντως οι εκλογές με το πιστόλι στον κορόταφο δεν γίνεται. Όλοι το λένε αυτό και, στον, και στην ΟΑΣΕ και στις δυτικές χώρες. Ε, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο του ΟΑΣΕ ε, να γίνονται εκλογές με τα τάγκ σε 100 μέτρα δίπλα ή 200 μέτρα δίπλα. Εδώ λοιπόν συμφωνούμε. Το όλο θέμα τώρα της επέκτασης των κυρώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί διότι οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο. Εάν δεν εφαρμοστεί αυτό το εργαλείο, ε, Ξέρετε, με την προπαγάνδα του ο Πούτιν έχει πει στο όλο τον κόσμο ότι η Ρωσία ε, περιστοιχίζεται από εχθρούς. Και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις είναι αυτές οι οποίες κάνουν το ρωσικό λαό να υποφέρει. Ε, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά βέβαια ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι αυτές που υποφέρουν. Όχι από τις ε, ε ευρωπαϊκές κυρώσεις αλλά από τα αντίμετρα που πήρε το Κρεμλίνο επιβάλλει κυρώσει η Ρωσία, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ρωσικής επίθεσης ε, και επιβάλλει κυρώσεις στη συνέχεια ε, η Ρωσία, αντίμετρα δηλαδή, επειδή η, Ρωσία, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά εφάρμοσε του διεθνείς κανόνες. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μα είπατε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. να δω λίγο τα ερωτήματα με τη σειρά για το θέμα του κυρίου Τσέτινα κατά, κατά πόσο υπάρχει σχέδιο Β κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Ε, αν ήταν θα το ξέραμε. Τα συμβαλόμενα μέρη, η Ρωσία, η Ουκρανία, ε, είναι προσιλωμένα στη Συμφωνία του Μίνσκ και βέβαια στο σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων αλλά και οι λοιποί εταίροι, οι Αμερικανοί το ίδιο κάνουν. Ε, το πραγματικό σχέδιο Β θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Ε, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες ε, δεν μπορούμε τώρα να ξαναγράψουμε τη συμφωνία του Μίνσκ ούτε να αλλάξουμε εντελώς το πλαίσιο. Δηλαδή θα ήταν μια πραγματική εγκατάλειψη. Και αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, μιας και θα υπήρχε κίνδυνος κλιμάκωσης στο Ντομπάς. είναι μια μεγάλη περιοχή. Έτσι, 17.000 ε, ε, χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα με αστάθεια ε, εκτός ελέγχου. Ήδη έχουμε πρακτικές ε, έτσι, εγκληματικότητας και μαφίας στην περιοχή, ε, μέσα στην Ευρώπη όλα αυτά. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει η συμφωνία. Δεν μπορούμε να τα καταλήψουμε σε καμιά περίπτωση αυτά. Και κάτι άλλο τώρα για τις εκλογές και την ασφάλεια. Ναι, βέβαια, για να λάβουν χώρα εκλογέ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνουν εκλογέ ε, στο παρόν, στην παρούσα κατάσταση όπου έχουμε ε, πυροβολισμού ε, με ελαφρύ και βαρύ οπλισμό. Χρειάζεται ασφάλεια για να μπορέσουν να λάβουν χώρα εκλογέ. Κάτι άλλο, το ερώτημα του κ. Ντεμεσμέικερ για την ε, για τις νάρκες και την αποναρκοθέτηση. Ε, μπορούμε να ε, προσπαθούμε να παρεύουμε, αλλά χρειαζόμαστε και ένα μέρη, χρειαζόμαστε τους χάρτες, δεν μπορούμε να στείλουμε ομάδες ε, για να βγάλουν τις νάρκες αν δεν υπάρχει ασφάλεια και δεν έχουμε χάρτες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα συμβαλόμενα μέρη, τους τα εμπλεκόμενα μέρη, διότι δεν έχει νόημα εμείς να βγάλουμε κάπου τις νάρκες και να τις βάλουν αυτοί κάπου αλλού. Ε, θα πρέπει λοιπόν να, τα βρούμε και με τις δύο πλευρές, άλλως δεν γίνεται. Αυτό που είπε και ο Στροβεσίτσιος ε, για τις ε, απαλωτριώσεις, ναι, είναι σημαντικό το θέμα αυτό για μας, το συζητάμε στις συζητήσεις στην Νόρμαντι και συχνά ζητούμε από τη Ρωσία να πιέσει τις, τις αποσχιστικές δυνάμεις διότι πρέπει να σταματήσει ο φαύλος με τα μέτρα και τα αντίμετρα και που έχει οδηγήσει ε, σε αυτήν την ενίσχυση ε, του μετόπου ουσιαστικά στον Ντομπάς ε, που καθυλώνει το μέτωπο και κόβει, κατακαιρματίζει το έδαφος, δεν ανοίγει το δρόμο για κάποια λύση και είναι βεβαίως αρνητικό και για τους τοπικούς πληθυσμούς που ξαφνικά είναι φυλακισμένοι σε διάφορα κομμάτια γης. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό για μας. Τώρα για τη μορφή που θα πάρει το φόρμα τέλο πάντων, δεν ξέρω, ρωτήστε τον κύριο Τίλερσον ε, τι πιστεύει ακριβώ. Εγώ τα είπα πριν. Ε, η δική μα πρακτική απέναντι στου Αμερικανού είναι ότι συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους ε, Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχουμε και εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση της παρούσας, του παρόντος πλαισίου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα τώρα, για τον υβριδικό πόλεμο. Ναι, η κυρία Χάρμς αναφέρθηκε στο θέμα της απόσυρσης, της απεμπλοκής. Ακούστε, όταν δημιουργούμε ζώνες απεμπλοκής, υπάρχουν ήδη έτσι δύο, πολύ περιορισμένες, αλλά υπάρχουν. Ε, πρέπει να υπάρχει μια παρουσία για να καλύψει το κενό αυτό και συνήθως, σύμφωνα με τη συμφωνία, η αποστολή παρατηρητών του, της ΟΑΣΕ του Άσε είναι που, έχει αυτό το ρόλο. Η κυρία Καλνίτα ρώτησε για τις εκλογές και την ασφάλεια, νομίζω απάντησα ήδη. Τώρα για τις κυρώσεις. Αυτό θα συζητηθεί βέβαια σε δύο μέρες ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διάρκεια των κυρώσεων σχετίζεται με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Αυτό θα εξετάσουν αύριο ε, μεθαύριο μάλλον η αρχηγοί κατών κυβερνήσεων. Ε, τι άλλο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ναι, ε, υπόθηκε ότι πρόκειται για μια σύραξη που είναι καθυλωμένη. Ναι, εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό βέβαια. Ε, ούτως ή άλλως ε, δεν, πρόκειται, δεν πρόκειται να παγώσει αυτή η σύραξη διότι είναι πολύ μεγάλη η κλίμακα των δυνάμεων που εμπλέκονται. Ε, από την τελευταία παρέμβασή μας, επειδή ρωτήθηκε τι έχει γίνει, τι νέο έχει συμβεί, ποιες είναι οι εξελίξεις, το πιο σημαντικό νομίζω είναι όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε. Μπορεί να μην είναι βέβαια τόσο ορατή και σε πολιτικό επίπεδο για τα διάφορα κείμενα, το πώς θα γίνουν εκλογές, ε, τα τέσσερα θεματικές, θεματικές τομείς, αλλά και για την ασφάλεια με τη διαπραγμάτευση ε, συμφωνιών τομεακών ε, για τα όπλα κάτω από 100 χιλιοστά, για την ε, εξάλληψη των αρκών. Όλα αυτά έχουν προχωρήσει, είναι έτοιμα, αλλά χρειάζεται πλέον πολιτική βούληση για να φτάσουμε στη τελική συμφωνία. Ναι, παρακαλώ, έχει μείνει ένα λεπτό. Ε, ε πολύ σύντομα, ε, κυρία Χάμς, σχετικά με το αν η τα, οι μεγάλες απειλές είναι η ε, απειλή για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό ακριβώς είναι το οποίο και μας σωθεί. Ε, είναι θέματα με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά, διότι αυτό είναι ε, το οποίο κάνει τόσο σημαντική τη συγκεκριμένη σύραξη για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να κάνουμε τα πάντα ε, για να μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο την συγκεκριμένη διαμάχη, όχι μονάχα για τους ανθρώπους εκεί πέρα. Ε, τώρα όσον αφορά το σχέδιο Β για το ε, Μίνσκ δεν υπάρχει ε, σχέδιο Β. Αυτά, οι, αυτές οι συμφωνίες είναι αυτό το οποίο έχουμε για την ώρα. Η ε, πρόοδος είναι πολύ αργή όμως ε, το Μίνσκ είναι αυτό το οποίο οποτεδήποτε έχουμε συζητήσεις για την κατάσταση είναι και το να υπάρξει μια αποκλιμάκωση της, της κατάστασης. Το συζητήσαμε αυτό τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου και επίσης ε, στο πλαίσιο του Μίνσκ μπορούμε να συζητήσουμε και για θέματα τα οποία αφορούν τη βελτίωση της κατάστασης για ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές όπως είναι για παράδειγμα ε, για την ε, ανθρωπιστική κατάσταση αλλά και την οικονομική κατάσταση ώστε να βελτιωθεί ε, η κατάσταση. Δεν έχουμε μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων υπερβολικές ε, προσδοκίες, όμως έχουμε την ρεαλιστική προσέγγιση των ε, μικρών βημάτων. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τους κατασμένους μας για τις δηλώσεις τους και τους συναδέλφους. Σε μερικά λεπτά θα ξεκινήσουμε αμέσως και με το επόμενο θέμα μας. Ευχαριστώ πολύ.